Καλημέρα σας, συνάδελφοι. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Μία πληροφορία καταρχήν να σας κοινοποιήσω δυνάμει του κανονισμού αποφάσισα κατά του Ιωάννη Λαγού, διότι στις 29 Ιανουαρίου 2020 ε, θορύβησε την Ολομέλεια χρησιμοποιώντας ε, λόγο ο οποίος δεν συνάδει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβάλλοντας και ε, συγκεκριμένο λεξιλόγιο, γι' αυτό για 7 ημέρες δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης και δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εργασίες του Κοινοβουλίου για τέσσερις ημέρες από σήμερα, 11 Φεβρουαρίου. Φυσικά η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής στο Προεδρείο Δυνάμει του Κανονισμού. Έχουν εγκριθεί τα πρακτικά της χτεσινής ε, συνεδρίασης, μάλλον έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις, δεν υπάρχουν, άρα εγκρίνονται τα πρακτικά της χτεσινής συνεδρίασης. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την έκθεση του κυρίου Μαυρίδη για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως προς την ετήσια έκθεση 2018. Δίνω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μαυρίδη και ε, χαιρετίζω και την κυρία Λαγκάρτ και τον Επίτροπο Ντομπρόφσκης. Κύριε Μαυρίδη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πηγαίνω κατευθείαν στην έκθεση. Η έκθεση αυτή αντικατοπτρίζει την ε, καλή σχέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βασικά είναι το βασικό εργαλείο σύμφωνα με το οποίο μπορούμε να εκφράσουμε απόψεις ε, για την σταθερότητα των τιμών, την ενίσχυση των οικονομιών της Ευρωζώνης και να οδηγήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό οικονομικής ε, Σύγκλησης. Η έκθεση αυτή είναι η πρώτη ε, του νέου νομοθε... της νέας νομοθετικής θητείας μετά την εκλογή της νέας Προέδρου της ΕΚΤ. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, χαιρόμαστε πολύ κυρία Λαγκάρτ που σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Η έκθεση έχει να κάνει με την αναθεώρηση των πρόσφατων πρακτικών ε, στην νομισματική πολιτική για την κλιματική αλλαγή και έναν πιο ισχυρό ρόλο ε, της Ευρώπης στον κόσμο για στα νομισματικά θέματα. Ε, μιλάμε συγκεκριμένα για την έκθεση της Κομισιόν του 2019 και ε, καλωσορίζουμε το ρόλο της ΕΚΤΕ στην νομισματική πολιτική και στη διασφάλιση της σταθερότητας ε, της οικονομίας. Οι προτάσεις τους οδήγησαν σε οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση των οικονομικών συνθήκων και την αύξηση των μειωμένων αποδόσεων σε πολλές τάξεις επενδύσεων. Τα επιτόκια δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές, τις εταιρείες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και όλους όσοι μπορούν να επωφεληθούν από, τη μεγαλύτερη, από το ρυθμό της οικονομίας, από τη μείωση της ανεργίας κτλ. Επίσης, ζητάμε από την ΕΚΤ να συνεχίσει να παρακολουθεί τους πιθανούς κινδύνους ε, ε, ως προς την πληθωρισμό των τιμών αλλά και τις επιπτώσεις ε, στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά συστήματα. Επίσης, ε, κρούμε τον κόδωνα ε, γιατί μετά από ένα μεγάλο διάστημα ανάπτυξης αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη έχουμε επιβράδυνση της ανάπτυξης από το 1,9% στο 1,1%. Επίσης, όσον αφορά το γεγονός ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να ε, διατηρηθεί μόνο μέσω της νομισματικής πολιτικής, υπογραμμίζουμε το ρόλο της δημοσιονομικής πολιτικής. Επίσης, ε, συμφωνούμε με τη δήλωση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι η αναθεώρηση του πλαισίου της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι κάτι που πρέπει να γίνει και χρειάζεται σε αυτή τη χρονική στιγμή. Θέλουμε να το ενισχύσουμε με δημόσια διαβούλευση και την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, το σημαντικό εδώ είναι το έβριμα ε, της ε, ομάδας των εμπειρογνωμόνων ε, της Eurostat που λέει ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της ανάκαμψης της αγοράς εργασίας και του μισθολογικού κόστου. Σύμφωνα με την έκθεση του Αυγούστου 2019, 6,2% ε, ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 7,4% στην Ευρωζώνη η ανεργία. Όμως αυτός ο ρυθμός δεν αντικατοπτρίστηκε στην αύξηση των μισθών. Επίσης για την ενίσχυση ε, του ρόλου της Ευρωζώνης. Χρειάζονται οι κατάλληλες ε, διαφορετικές συνθήκες εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής Ένωσης, ε, η ε, εξασφάλιση των καταθέσεων. Επίσης δίνεται έμφαση στην πάταξη της κλιματικής αλλαγής και την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων. Επίσης, η ΕΚΤ δεσμεύεται από την Συμφωνία του Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και από τις αρχές σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό και επίπεδο διακυβέρνησης. Όσον αφορά το Brexit, ε, την ε, Ένωση Κεφαλαγορών, τα κρυπτονομίσματα, το ρυθμιστικό πλαίσιο, την σημασία των μικρών, πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την πρόσβαση στις πιστώσεις, θεωρούμε ότι ε, πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο για να ενισχυθεί και η πραγματικότητα πραγματική οικονομία. Ως προς τη λογοδοσία, υπό την Προεδρία του Μάριο Ντράκη είδαμε αύξηση της λογοδοσίας και ελπίζουμε και προφράζουμε τη βούλησή μας για μεγαλύτερο διάλογο, λογοδοσία και ανοιχτή τη σχέση και με την ε, τωρινή πρόεδρο. Επίση είναι σημαντικό όχι μόνο να διαμορφώνουμε νομισματικές πολιτικέ, αλλά να τι επικοινωνούμε και προ του πολίτε, οι οποίοι πρέπει να κατανοούν τον αντίκτυπο που έχουν αυτέ στη ζωή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του σκιώδε εισηγητέ για την επικοδομητική συνεργασία τους ε, και να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ΕΚΤ έχουν έναν κοινό στόχο και αυτό ήταν και για μένα ο πρωταρχικό στόχο όταν συνέταξα αυτή την έκθεση, να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών μας επιτυγχάνοντας πραγματική οικονομική σύγκληση και να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς είναι το κοινό μας σπίτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Μαυρίδη. Τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Κριστίν Λαγκάρτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Σιγητά, κύριε Μαυρίδη, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω για πρώτη φορά σε μια ολομέλεια εδώ και να συζητήσω το σχέδιο εκθεσή σα όσον αφορά την ετήσια έκθεση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το έτο 2018. Η ανεξαρτησία και η λογοδεσία αποτελούν δύο πλευρέ του ίδιου νομίσματο για την ΕΚΤ και το ένα δεν μπορεί να υπάρχει χωρί το άλλο. Και γι' αυτό ακριβώς η σχέση της ΕΚΤ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τόσο σημαντική. Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της σχέσης αυτής και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον καλό διάλογο που έχουμε μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων μας. Βρέθηκα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από 100 μέρες, σχεδόν ακριβώς. Διαβάζω την έκθεση αυτή με πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι ακριβώ εκτιμάμε με τον ίδιο τρόπο τις προκλήσεις, πολλέ από τι προκλήσει που αντιμετωπίζει τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και η Ευρωζώνη. Και αισθάνομαι ακριβώ το ίδιο όπως και εσείς κύριε Σιγητά, τώρα που σα άκουγα. Πράγματι, η οικονομική φύση των προκλήσεων απαιτούν συνεχή διάλογο μεταξύ μας. Και σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο κυρίως ε, προκλήσεις και ανησυχίες που αναφέρονται στην έκθεσή σας. Πρώτον, ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον και δεύτερον, οι διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία της Ευρωζώνης σήμερα. Η Ευρωζώνη και η ανάπτυξή της και ο ρυθμό μάλλον ανάπτυξης έχει επιβραδυνθεί από τι αρχές του 2018 κυρίω εξαιτία παντακοσμίων αβεβαιοτήτων και αδυναμιών στο διεθνέ εμπόριο. Ο έλεγχος της ανάπτυξης αυτής που είναι όντως μειωμένη έχει επηρεάσει τις τιμές και ο πληθωρισμός παραμένει κάτω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας. Συνεπώς, στα πλαίσια αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έδρασε με αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να πετύχει τη σταθερότητα των τιμών που είναι και η εντολή η οποία έχουμε εμείς βάσει της συνθήκης. Η νομισματική μας πολιτική από το 2014 βασίζεται σε τέσσερα στοιχεία. Από το 2014, έτσι. Αρνητικά επιτόκια, αγορές ενεργητικού, ενδείξεις και δραστηριότητες δανεισμού. Αυτά τα μέτρα έχουν βοηθήσει προκειμένου να πετύχουμε ευνοϊκέ συνθήκες δανεισμού, να στηρίξουμε την αντοχή της εσωτερικής οικονομίας και κυρίως, κυρίως πρόσφατα να προστατεύσουμε την οικονομία της Ευρωζώνης από δυσκολίες στο διεθνές επίπεδο. Η πολιτική μας λοιπόν έχει στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη που οδήγησε σε περισσότερες θέσεις απασχόλησης και σε υψηλότερους μισθούς για τους πολίτες της Ευρωζώνης. Όπως ήδη αναφέρατε κύριε Σιγητά, η ανεργία στην Ευρωζώνη, 7,4% είναι στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2008. Οι μισθοί, επίσης αναφερθήκατε και στους μισθούς, αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 2,5%. Τα πρώτα τρία τετράμινα του 2019, πάνω δηλαδή από το μέσο όρο μακροπρόθεσμα. 2,5%. Όμως η νομισματική πολιτική δεν μπορεί και ούτε πρέπει να είναι το μόνο, ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει τα πράγματα. Όσο πιο πολύ κρατούν τα διευκολυντικά μας μέτρα, τόσο περισσότερο ελοχεύει ο κίνδυνος παρενεργειών, που θα γίνουν όλο και περισσότερο έντονες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων επηρεάζει ε, τα έσοδα από τις αποταμιεύσεις, ότι ολοχεύουν κίνδυνοι και στις ε, τιμές της κατοικίας. Παρακολουθούμε λοιπόν τις αρνητικές παρενέργειες έτσι ώστε αυτές να μην βαρύνουν υπερβολικά ε, τις θετικές επιπτώσεις των μέτρων που υιοθετούμε για την πιστοτική δραστηριότητα είτε τους μισθούς, είτε τα των οικοκυριών. Για παράδειγμα, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισάγει ένα νέο μέτρο για να ε, από ουσιαστικά για να βοηθήσει τις ε, τράπεζες εκείνες οι οποίες έχουν αρκετά κεφάλαια στη διάθεσή τους. Άλλα μέτρα επίσης, όπως τα δημοσιονομικά μέτρα, όπως διαρθρωτικές πολιτικές, επίσης μπορούν να παίξουν το δικό τους ρόλο. Οι πολιτικές αυτές μπορούν να ενισχύσουν την αύξηση της παραγωγικότητας και να βοηθήσουν και το δυναμικό ε, της Ευρωζώνης. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τα μέτρα μας. Όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά, η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να είναι αποτελεσματική, μπορεί να στηρίξει τον ρυθμό ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και να ενισχύσει την βοήθεια στην πίεση που δέχονται οι τιμές και να αυξηθούν έτσι τα επιτόκια σιγά σιγά. Η Πράσινη Συμφωνία η πρωτοβουλία για την οικολογική μετάβαση επίσης μπορούν να βοηθήσουν συνεισφέροντας σε μεγαλύτερη ανάπτυξη. οικονομική ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το σχέδιο έκθεση για την ετήσια έκθεση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφέρεται σε τρει διαρθρωτικέ εξελίξει που επηρεάζουν το οικονομικό μας περιβάλλον. Το ένα είναι η ψηφιοποίηση, το άλλο είναι η κλιματική αλλαγή και το τρίτο είναι η θεσμική αρχιτεκτονική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Και θα ήθελα εδώ να χρησιμοποιήσω το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου για να συζητήσω μαζί σας αυτές τις τρεις προκλήσεις. Η ψηφιοποίηση και η κλιματική αλλαγή είναι πράγματα τα οποία δεν έρχονται από την Ευρώπη μόνο, είναι παγκόσμια φαινόμενα και δεν θα μας περιμένουν να προετοιμαστούμε για να τα αντιμετωπίσουμε. Θα μας επηρεάσουν, είτε είμαστε έτοιμοι είτε δεν είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει τις δυνατότητες και τις επιπτώσεις των τεχνολογικών εξελίξεων για τις πληρωμές και για την σταθερότητα των τιμών. Και επίσης συνεισφέρει σε τέτοιου είδους καινοτομίες. Εξού και έχουμε δημιουργήσει μία task force στο ευρωσύστημα από τον Ιανουάριο ώστε να εξετάσουν τις προκλήσεις και τον σχεδιασμό που μπορούμε να έχουμε για κρυπτονομίσματα και πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο να λειτουργήσει στην πράξη. Επίσης θέλουμε να εκτιμήσουμε κατά πόσο ένα ψηφιακό νόμισμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα μπορούσε να βοηθήσει το κοινό και να στηρίξει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μαζί λοιπόν με πέντε άλλες κεντρικές τράπεζες και με την Τράπεζα Διακανονισμών θα ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες και θα εκτιμήσουμε την χρησιμότητα διασυνοριακά ενός τέτοιου ψηφιακού νομίσματος. Επίσης, πρέπει να επιταχύνουμε και όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και όχι μόνο γιατί μας νοιάζει επειδή είμαστε πολίτες του κόσμου. Η ψηφιοποίηση αλλά και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι κεντρικές τράπεζες. Οπότε θέλουμε όλο και περισσότερο να λάβουμε υπόψη μα αυτές τις παραμέτρους στις πολιτικέ μας και στις δράσεις μας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτον, εργαζόμαστε για να μάθουμε περισσότερα όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και να διασφαλίσουμε ότι οι επιπτώσεις της αντικατοπτρίζονται στις οικονομικές μας αναλύσεις, στις προβλέψεις που κάνουμε και στη μεθοδολογία μας. Δεύτερον, μέσω των ε, καθηκόντων τη που είναι η σταθερότητα των τιμών εξετάζει του συστημικού κινδύνου που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και τι προσπάθειε επίση για να έχουμε μια οικονομία χωρί άνθρακα. Έτσι μπορούμε να δοκιμάσουμε και να δούμε πόσο καλά ο τραπεζικός τομέας της Ευρωζώνης μπορεί να αντιμετωπίσει κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Και τέλος, η ΕΚΤ έχει αναλάβει βήματα ώστε να ευθυγραμμίσει τις δικές της αποφάσεις για επενδύσεις ε, σύμφωνα με την Συμφωνία των Παρισίων για παράδειγμα το συνταξιδοτικό ταμείο του προσωπικού μας και αποφασίσαμε να πάμε σε άλλο δίκτυο, χαμηλότερου άνθρακα και προσπαθούμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στις δράσεις μας στις αγορές. Έπειτα υπάρχει και η επανεξέταση της στρατηγικής μας, η οποία βασίζεται στις τόσο γρήγορες αλλαγές που έχουμε στα ψηφιακά, στη βιωσιμότητα και στην παγκοσμιοποίηση όπου εμπλέκονται βέβαια οικονομικές δαμές και να δούμε πώς αλλάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η νομισματική πολιτική. Αυτή η επανεξέταση της στρατηγικής μας θα εξετάσει όλες τις πτυχές του πλαισίου πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να φέρουμε σε πέρα την εντολή μα που είναι σταθερότητα των τιμών προ όφελο όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Μέρος τη διαδικασία αυτή θα είναι διαβούλευση με το κοινό και θα ακούσουμε τις απόψει τους, τις προσδοκίες τους και τις ανησυχίες τους. Και αυτό με ανοιχτό πνεύμα. Πράγματι, θα συνεργαστούμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όσους από εσά εδώ ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για αυτά τα ζητήματα, κάτι το οποίο έχουμε ήδη ξεκινήσει. Τώρα, Έχω επικεντρωθεί μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι όμω σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η ψηφιοποίηση και η κλιματική αλλαγή αποτελούν οικουμενικέ εξελίξει που μα επηρεάζουν όλου, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά παντού. Η Ευρώπη βέβαια βρίσκεται σε μια ειδική θέση για να αντιμετωπίσει τι προκλήσει αυτέ. Μπορεί να χτίσει πάνω σε κίνητρα, ε, πάνω σε ό,τι μα προσφέρει η ενιαία αγορά που προσφέρει πολλά για τον εξυγχρονισμό τη αγοράς μας και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε σωστές απαντήσεις στις προκλήσεις που μας περιμένουν. Όμως, πρέπει να ξέρουμε ότι ένα σημαντικό πυλώνα τη απάντηση της Ευρώπης σε ένα κόσμο που παγκοσμιοποιείται όλο και περισσότερο, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση δεν πρέπει να ξεχαστεί. Και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι συνομοθέτης μπορεί να βοηθήσει να έχουμε τη σωστή απάντηση. Μην υποτιμάμε αυτό το ρόλο. Η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης έχει εξελιχθεί. Όπως όμως γνωρίζετε, κάποια βασικά στοιχεία εξακολουθούν να λείπουν ή δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πρέπει να μπορεί να προσφέρει στο ύψος των δυνατοτήτων που έχει το σύστημά μας. Εξού και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητάει και θα συνεχίσει να το κάνει μια περισσότερο ολοκληρωμένη οικονομική και νομισματική ένωση. Και οικονομική και νομισματική. Πολύ σύντομα τώρα επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω τι εννοώ με αυτά. Πρόκειται για μια πλήρη τραπεζική ένωση. Πρόκειται επίση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων. Πρόκειται για μια πραγματική ένωση κεφαλαίου αγορών με καινοτομία και με λειτουργία σταθεροποίηση προκειμένου να μπορούμε να προστατευτούμε όταν αυτό χρειάζεται. Επίσης, μια οικονομική και νομισματική ένωση με περισσότερη αντοχή που θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε τα επίπεδα ζωής μας μέσα στις διάφορες εξελίξεις, αλλά θα στηρίξει και την επιρροή της Ευρώπης ανά το κόσμο και θα φροντίσει το ευρώ να είναι πιο να προσελκύει περισσότερο κόσμο και να χρησιμοποιείται ευρύτερα. Και θα ολοκληρώσω αναφερόμενοι στις κοινέ προκλήσεις. Αυτά τα οποία συζητάμε τώρα τι σημαίνουν. Σημαίνουν ότι όλοι πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν, όσο περισσότερο μπορούν. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βέβαια, η οποία στα πλαίσια τη εντολή τη είναι έτοιμη να παίξει το δικό τη ρόλο. Και όπω είπα στην αρχή, ο οικουμενικό χαρακτήρα των προκλήσεων αυτών έχει σαν αποτέλεσμα να πρέπει να συνεχιστεί επιμονή μου βάση ο διάλογο ανάμεσα ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσβλέπω λοιπόν στην ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε μεταξύ μα ε, σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ την πρόεδρο Λαγκάρτα. Ε, κύριε Ντομπρόφσκης, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχετε το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητή Πρόεδρε της ΕΚΤ, αγαπητά μέλη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συζητήσουμε σήμερα για την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ ε, έχει ξεκινήσει με μία αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΚΤ ε, για, ήδη τον Ιανουάριο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κώστα Μαυρίδη και την ε, Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Σημεριζόμαστε τις θέσεις ε, της έκθεσης σε γενικές γραμμές. Αυτό που έχει σημασία είναι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ ε, ως προς την νομισματική πολιτική για να ενισχύσει την νομισματική σταθερότητα. Αυτό αφορά και τις διαδικασίες δημοκρατίας και λογοδοσίας. Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ δεν αρκεί για την βιώσιμη ανάπτυξη και σταθερότητα των τιμών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ένα μείγμα διαρθρωτικών πολιτικών και προσαρμογή της χρηματοοικονομικής πολιτικής. Αυτό είναι ύψης της σημασίας για την ανάπτυξη της οικονομίας τη στιγμή που υπάρχει χαμηλότερος ε, ρυθμός ανάπτυξης με βάση και τις ολισθήσεις που υπάρχουν στις εμπορικές πολιτικές. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά σημεία της έκθεσης που σχετίζονται με την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει προτεραιότητα στις κλιματικές αλλαγές και τα περιβαλλοντικά και γι' αυτό ακριβώς θα υπάρχει μία τυποποίηση και καινοτομία καθώς και ένας διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και διεθνής συνεργασίας. Μέσα στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας συμφωνούμε με τα συμπεράσματα της ΕΚΤ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους ε, κινδύνους των κλιματικών αλλαγών που θα γίνουν πιο συστημικοί αν δεν γίνουν οι δέουσες αλλαγές. Επίσης, ως προς την βιώσιμη χρηματοοικονομική πολιτική και χρηματοδότηση, η πολιτική μας θα δημοσιοποιηθεί στις αρχές του φθινοπόρου έτσι ώστε να ενταχθούν αυτά τα δεδομένα στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Επίσης θα ορίσουμε μία τυποποίηση των πρασίνων ομολογιών ως προς τις μελλοντικές επενδύσεις. Επίσης και εμείς θα λάβουμε υπόψη μία αναθεώρηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη την βιωσιμότητα της οικονομίας που αποτελεί όρο ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Θα πρέπει όμως να είμαι πιο αποδοτικοί. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αγορά, η ένωση μάλλον κεφαλαιαγορών, με βάση και το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Έτσι ενθαρρύνουμε το Κοινοβούλιο να συνεργαστεί με την ΕΚΤ και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εμείς έχουμε αρχίσει τις ε, τεχνικές εργασίες για την αντιμετώπιση κρίσεων και το νομοθετικό πλαίσιο περί για να γίνει μία ε, πρόοδος ως προς την Τραπεζική Ένωση. Έχει μεγάλη ε, σημασία η έργασή μας και για τις πληρωμές και τα κρυπτονομίσματα. Ευχαριστώ πολύ την ΕΚΤ για την εργασία της ως προς τις ε, διαρθρώσεις και τη δομή άμεσων πληρωμών ενδοευρωπαϊκά και αυτό αφορά και, την, ε, και τις ψηφιακές πληρωμές έτσι ώστε οι πληρωμές να μην γίνονται και να μην είναι τόσο δαπανηρές. Είμαι πεπισμένος ότι η σημερινή συζήτηση θα είναι ιδιαίτερα επικοδομητική και θα υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ ΕΕΚΤ και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας ακούσουμε τώρα τις πολιτικές ομάδες. Από το ΕΛΚ ο κύριος Φέρμπερ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Είναι αρκετά καλά τα γερμανικά σας, κυρία Λαγκάρτ, λιγάκι, ε. Ευχαριστώ. Ε, καταρχάς που ήρθατε σήμερα εδώ για πρώτη φορά ε, υπό τη νέα σας ε, ε, θέση ως ε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εμείς στην ε, Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή σας εγγυόμαστε ότι θα φροντίσουμε για τη σταθερότητα του νομίσματος που είναι η εντολή σα, αλλά ότι θα συνεχίσουμε και το διάλογο με τον κοινό προς το ρόλο που έχει να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Ο προκάτοχός σας, ο οποίος ερχόταν σε εμά τακτικά με τα μέτρα του στην νομισματική πολιτική, συνέβαλε ώστε να αγοράσουμε χρόνο ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να τον χρησιμοποιήσουν ε, ε, σε κάθε πλευρά και για την προετοιμασία για δύσκολους καιρούς. Ε, εσείς αναγγείλατε μια νέα πολιτική για την οποία θα ήταν καλό να συζητήσουμε. Ελπίζουμε η φάση κατά την οποία υπάρχουν εσωτερικές συζητήσεις στην ΕΚΤ να μην μπει στον πάγο, να μπορέσουμε να αντιδράσουμε έγκαιρα έτσι ώστε να δούμε τη σειρά των προβλημάτων ε, τα οποία μπορεί να προκύψουν όταν έχουμε μια τέτοια μακρά φάση και έχουμε χαμηλούς ε, ε, τόκους που στην ουσία οδηγούν σε αυτά τα προβλήματα. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε την ψηφιακή εποχή και τα ψηφιακά νομίσματα. Είναι καλύτερα να έχουμε ένα ψηφιακό νόμισμα από την ΕΚΤ παρά από το Facebook. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο ε, Φέρμπερ. Ο επόμενος που ζήτησε το λόγο είναι ο κύριο Φερνάντε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ το νέο αυτό αέρα που έχει φέρει η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ στο Σώμα και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά θέλω να επιμείνω επίση και για το ότι ακόμα είμαστε μακριά από το να έχουμε τηρήσει την εντολή στα νομισματικά, στη πιστοτική διάσταση. Χρειάζεται γρήγορα να προχωρήσουμε και να φέρουμε τον πληθωρισμό κοντά στο 2%. Οπότε, στα πλαίσια τη ανεξαρτησία ε, βέβαια του θεσμικού σα οργάνου, θέλω να επιμείνω ότι χρειάζονται νέα μέσα, νέε πολιτικέ για να μπορέσουμε τον πληθωρισμό να τον πάμε κοντά στο στόχο του. Έπειτα, θέλω επίσης να σας συστήσω να ζητήσετε πραγματικά στήριξη στο δημοσιονομικό σκέλος για να μπορέσετε εσείς να πετύχετε το στόχο σας. Και σε αυτήν την επανεξέταση της στρατηγικής σας δεν θα πρέπει απλώς να αλλάξετε λιγάκι τη μεθοδολογία, αλλά να εισάγετε νέους στόχους, νέα μέσα, όπως θέλετε πείτε το, στο έργο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος Λουίς Καρικάνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντομπρόφσκη. Καλώ ήρθατε κύριε Λαγκάρτ. Πολύ χαίρομαι που σα βλέπω εδώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κύριο Μαυρίδη για το εξαίρετο έργο του όσον αφορά την έκθεση αυτή. Όπως βλέπετε και στην έκθεση κυρία Λαγκάρτ, εμείς ανησυχούμε που δεν έχει ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Και χαίρομαι που άκουσα τον κύριο Ντομπρόφσκης να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα εργασία τη θα πιέσει προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Χαιρόμαστε επίση για αυτά που σας ακούσαμε να λέτε για τις προτεραιότητές σας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Πιστεύουμε ότι αν υπάρξει άλλη τέτοια κρίση, τότε έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα δεν θα φτάσει. Κανονικά πρέπει να αποτελούνται από τρεις πυλώνες το έργο μας. Τώρα έχουμε τους δύο πυλώνες, ο τρίτος πυλώνας, η εξυγίανση πραγματικά δεν εφαρμόζεται ακριβώς. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, αλλά πάντως δεν φτάνει για να λυθούν ε, πολλές περιπτώσεις τραπεζών σε περίπτωση που χρειαστεί. Και βέβαια ο τρίτος πυλώνας εννοείται η εξασφάλιση καταθέσεων δεν έχει προχωρήσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια τραπεζική ένωση η οποία να κόψει ε, την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις τράπεζες και τα κράτη. Δεν πρέπει τα κράτη να διασώζουν τις τράπεζες. Άρα η Επιτροπή έχει πολλά να κάνει ακόμα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάντως να ξέρετε ότι εμείς σας στηρίζουμε και ζητάω την στήριξη και της κυρίας Λαγκάρτ βέβαια και του Αντιπρόεδρου Ντομπρόφσκης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος στον κύριο ε, Γκούναρ Μπέκε. Ευχαριστώ την κυρία ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με αυτή την ετήσια έκθεση ε, αυτό το ε, έφυγε ο Μάριο Ντράγκη από αυτό εδώ το σώμα. Μίλησε για την ανάπτυξη και πραγματικά ο Ντράγκη είχε ασκήσει τη μεγαλύτερη πίεση ε, από οποιονδήποτε άλλο στα νομίσματα από το 1925. Είδαμε στην Bank of England ε, να αυξάνονται οι ε, τόκοι. Είδαμε ότι ο Τράγκη δεν χρησιμοποιούσε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το 2009 ήμασταν σε μεγαλύτερη θέση από ότι η αμερικανική οικονομία, οικονομία και η κρίση μας χτύπησε πολύ δυνατά. Το 2018 ο Ντράγκη ε, ε, έδωσε στην Ευρώπη περισσότερους ανθρώπους αλλά μικρότερη οικονομία. 35% μείωση είχαμε. Πραγματικά πόσο μεγάλες οι επιπτώσεις στους νέους. Στην ε, Γερμανία λιώνουν οι ηλικιωμένοι γυροκομεία όπως λιώνουν οι πάγοι στην Ανταρκτική. Έχουμε επίσης αύξηση της ε, περιουσίας ε, των ε, ανθρώπων με μεγάλο πλούτο στα χέρια τους. Επίσης με την πολιτική αρνητικών επιτοκίων του Τράγκη δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την φαντασία σου του για την οικονομία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιάκελ Γιούνιας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Μαυρίδη, ο οποίος ε, οδήγησε σε μία έκθεση σύγκλησης θέσεων όλων των πολιτικών ομάδων για την γενική μας θεώρηση ως προς το μέλλον της ΕΚΤ. Κύριε Λαγκάρντα, όταν, σας, ε, όταν ε, ζητήσαμε τη γνώμη σας για τα ψηφιακά νομίσματα στην ακρόασή σας, είπατε ότι θα δράσετε, αλλά όχι με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έχετε κατανοήσει βεβαίως ε, το θέμα και τη σπουδή με την οποία θέλουμε να το προωθήσουμε. Επίσης, θα πρέπει να γίνει μία συζήτηση για την, ε, για το τομέα της ε, επιθεώρησης και του ελέγχου του χρηματοοικονομικού τομέα, γιατί ε, δυστυχώς είναι μεν σαφείς οι εντολές όλων των οργάνων, αλλά ως προς την Ένωση των Κεφαλαιαγορών και την Ένωση των Τραπεζών βλέπουμε ότι ε, δεν ακολουθούν το ρυθμό που θα θέλαμε. Χρειάζεται λοιπόν μια νέα δυναμική για αυτούς τους δύο τομείς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θέλαμε να δώσετε μια νέα πνοή σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε ο κύριος Φανόφερτφελτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η σταθερότητα των τιμών είναι ο πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ. Δεν μπορείτε να έχετε σταθερότητα τιμών χωρίς χρηματοοικονομική σταθερότητα που αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα τιμών. Τι βλέπουμε όμως στην Ευρώπη, χαμηλά επιτόκια, σπρέντ ε, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σωστά, συγχωνεύσεις, κερδοσκοπίες, ε, σκιώδεις τραπεζικής, τραπεζικές δραστηριότητες και 15-3 δολάρια αρνητικών αποδόσεων. Μπορούμε να πούμε, αν δείτε αυτές τις εξελίξεις, ότι δυστυχώς η χρηματοοικονομική σταθερότητα δεν υφίσταται. Επίσης, η, η μη συστημικές οικονομικές πολιτικές είναι αυτές που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Παπαδημούλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Λαγκάρτ, σας καλωσορίζουμε στην Ολομέλη, όπως και σας κύριε Ντομπρόφσκης. Αλλά νομίζω ότι ο μεγάλος ένοχος για αυτά που κάνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανησυχεί είναι απόν από αυτή τη συζήτηση και το μεγάλο φρένο σε αυτά που πρέπει να κάνουμε είναι το συμβούλιο είναι οι κυβερνήσει. εκεί μπλοκάρει η ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης και ο τρίτος πυλώνας κύριε καρικάνο. στο συμβούλιο γιατί η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα ζητάει το έντι. η κομισιόν το προτείνει στο ευρωκοινοβούλιο η πλειοψηφία το θέλει. και ο κίνδυνο δεν είναι μόνο η οικονομική επιβράδυνση ο κίνδυνο είναι μια νέα οικονομική κρίση κυρία λαγκάρντ και δέκα χρόνια μετά την κρίση που ξέσπασε στις ηνωμένες πολιτείες οι ηνωμένες πολιτείες έχουν ανακάμψει και εμείς ακόμη συζητάμε το πλαίσιο το ενισχυμένο της οικονομικής διακυβέρνησης που θα βαθύνει την πολιτική την οικονομική την νομισματική ενοποίηση και θα καταστήσει την ευρωπαϊκή ένωση και την ευρωζώνη πιο ισχυρή. και αυτό λείπει. όπως λείπουν και τα χρηματοδοτικά μέσα για να υλοποιηθεί το green deal διότι και πάλι το συμβούλιο θέλει να περικόψει τον οικονομικό προϋπολογισμό για το νέο πολιετές πλαίσιο σε αντίθεση με το ευρωκοινοβούλιο που ζητάει περισσότερα χρήματα για να μειωθούν οι ανισότητες για να επενδύσουμε στην αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης για να κρατήσουμε την πολιτική συνοχή για να φύγουμε μπροστά με επενδύσεις στην καινοτομία. επομένως η έκθεση του κ. μαυρίδη είναι μια ευκαιρία για να δούμε τι πρέπει να αλλάξει για να συμπαρασύρουμε και αυτούς που βάζουν φρένο. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο, ο κύριος Μάρτο Κυρανγκιουσί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως πολύ σωστά τονίζει η έκθεση, το ευρώ δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο οικονομικό ή νομισματικό, είναι και συμβολικό. Και αν θέλουμε το ευρώ να αποτελέσει αποθεματικό νόμισμα, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του προβλήματος και των αδυναμιών που αναφέρει ακριβώς η έκθεση. Η μακροπρόθεσμη σταθερότητα του ευρώ ω νόμισμα εξαρτάται από το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να αντιμετωπίσει τι γεωγραφικέ διαφορέ και τι διαρθρωτικέ επίση αλλαγέ που παραμένουν και διαφορέ που παραμένουν μεταξύ των χωρών μελών και που εκφράζονται σε διαφορές μισθών ανάμεσα στις παλιές και τις νέες χώρες μέλη, για παράδειγμα. Αυτές οι ανισορροπίες έχουν πολύ σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, όχι μόνο στην ανταγωνιστικότητα, αλλά και στην ανεργία των νέων, όπως επίσης και στην μετανάστευση για να βρει δουλειά ε, κανείς αλλού. Και όπως πολύ σωστά λέτε κυρία Πρόεδρε, δεν χρειάζονται μόνο νομισματικά μέσα, αλλά και δημοσιονομικά. Η πολιτική συνοχής επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη, κατά πολέμηση της διαφθοράς Επίσης, προκειμένου να σταματήσει αυτή η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους μισθούς της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πιετικάινεν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω από βάθους καρδίες και να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη νέα της ηγεσία που επιτέλους θα έλεγα ε, παίρνει υπόψη της ε, ε, τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή ή λαμβάνει υπόψη τους περιβαλλοντικούς κινδύνους αλλά και τους συστημικούς κινδύνους τους τωρινούς και τους μελλοντικούς. Χαίρομαι λοιπόν που ακούω ότι όλα αυτά θα τα επανεξετάσετε στα πλαίσια της στρατηγικής σας και προσβλέπω στην επανεξέταση αυτή. Ελπίζω επίσης να υπάρξει και συνέχεια σε όλες τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο μέλλον και να χρησιμοποιηθούν ε, διάφορα μέτρα προκειμένου να μην χρηματοδοτούνται δράσεις, για παράδειγμα, που καταστρέφουν το περιβάλλον. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει βέβαια γρήγορα με το δικό της χρηματοδοτικό πακέτο και να λάβει υπόψη διάφορους παράγοντες. Σας παρακαλώ, λάβετε υπόψη σας ότι η δείκτες, η ανάλυση του κύκλου ζωής είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται και να ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία ε, στα διάφορα θεσμικά όργανα, ώστε πραγματικά να ξέρουμε τι κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, λίγο για πειθαρχία χρόνου ζητώ. Η πρόεδρος της ε, Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, η κυρία Τινάκλη. Άκρο, please, madame. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράζει την υποστήριξη των πολιτικών του, της ΕΚΤ και αναγνωρίζει την εντολή αυτή που συμβαδίζει ε, με τους στόχους στην Ευρωζώνη ως προς το αποπληθωρισμό και την οικονομική εξυγίανση. Θα ήθελα να μου πείτε αν πραγματικά φτάνουμε σε τέτοιους στόχους. Σας προκαλώ να μου το αποδείξετε. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς ορίζεται η νομισματική πολιτική. Μιλήσατε για τις κλιματικές αλλαγές, για την ψηφιοποίηση, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις οικονομικές ανισότητες, ιδιαίτερα σε ορισμένους τομείς. Αυτό θα δράσει ανελέητα κατά συγκεκριμένων τομέων. Θα πρέπει λοιπόν να φτάσετε σε σταθερότητα τιμών, αλλά για να το ε, φτάσετε αυτό θα πρέπει να κατανοήσετε καλύτερα τις κλιματικές αλλαγές που θα πλήξουν ε, τα νοικοκυριά, της ε, επιχειρήσεις και τα θεσμικά όργανα. Θα, εμείς τουλάχιστον θα ανταποκριθούμε ως προς το δικό μας ρόλο. Ευχαριστώ κυρία Στεφανίγιον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε που ήρθατε. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά για την εξεντρική σα έκθεση. Όπω και εσεί και εμεί συμφωνούμε με τη διαπίστωση αυτή για μια οικονομική ανάπτυξη ε, αδύναμη και ότι κάτι πρέπει να γίνει για την οικονομία μα. Εκπροσωπούμε του Ευρωπαίου πολίτε και εμεί διαπιστώνουμε τι ανησυχίε που έχουν επιτόπου, γιατί αυτή η αδύναμη ανάπτυξη δεν βοηθάει ούτε την κατανάλωση, ούτε τις τιμές, ούτε και τις ε, τιμές ε, τη κατοικία που δεν είναι προσθέσει σήμερα. Έπειτα, η κατάσταση στην Κίνα, το Brexit, κινδυνεύουν να επηρεάσουν ακόμα περισσότερο την οικονομία μα. Αυτή λοιπόν την περίοδο αβεβαιότητα και ψηφιακή και οικολογική μετάβαση, χαίρομαι για την πρωτοβουλία σα, επανεξέταση στη στρατηγική σα τη νομισματική πολιτική, δηλαδή τη ΕΚΤ, που θα λάβει υπόψη όλε αυτέ τι αλλαγέ. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα, πολλά μέτωπα ανοιχτά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να κάνει πολλά για να έχουμε πραγματικά πρόοδο όσον αφορά την ισορροπία ανδρών γυναικών, στι ε, υψηλέ ε, θέσει ευθύνη στην ΕΚΤ. Αλλά επίση να παρακολουθήσουμε τι γίνεται και με τα κρυπτονομίσματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα ακόμα την νομοποίηση ε, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να ενισχύσουμε τον αποθεματικό ρόλο του ευρώ διεθνώς κλπ. Στην εκπόνηση της στρατηγικής αυτής χαίρομαι για την μεθοδολογία που προτείνεται ε, ανοίγματο και διαλόγου μαζί μας και είναι κάτι με το οποίο δεσμευτήκατε στην πρώτη σας ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι επίσης και για τη συνέχεια που θα δώσετε το Μάρτιο που θα έρθετε και θα μιλήσετε με την κοινωνία των πολιτών στις Βρυξέλλες και ελπίζω να συμμετάσχουμε και εμείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Λαπόρτ. Ε, κυρία Λαπόρτ. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε και που προσπαθείτε να συμβάσετε τα συμβαστά. Ε, πράγματι, θα δοκιμαστούμε πολύ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάνω απ' όλα, γιατί η συνέχεια τη Ευρωπαϊκή Νομισματική Πολιτική είναι σαν να γυρνάμε γύρω-γύρω, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό και την ανεργία. Ο κύριο Ντράγκη, ο προκάτοχό σα, ε, ε, και κατέβασε ακόμα περισσότερο τα επιτόκια και ακολούθησε μη συμβατικά μέτρα. Τα αρνητικά επιτόκια όμως αυτό που κάνουν είναι ότι πλήττουν τους αποταμιευτές και οδηγούν σε κερδοσκοπία. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια πιο κανονική κατάσταση και πώ εσεί θα βγείτε από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί η ΕΚΤ σήμερα. Έπειτα, ε, παρόλο που μιλάτε για την ανεξαρτησία τη ΕΚΤ, εσεί δηλώσατε ότι την κλιματική αλλαγή θα την καταστήσετε προτεραιότητα για να ανταποκριθείτε σε αυτά που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερο πράσινε επενδύσει, δηλαδή, αλλά εγώ θα έλεγα και περισσότερο πολιτικοποιημένε. Μια τέτοια κατάσταση όμω σημαίνει ότι ξεφεύγετε από την εντολή σα, τη στιγμή που αναλαμβάνετε τέτοιε αρμοδιότητε και είναι και σε βάρος τη κυριαρχία των χωρών μελών. Πώ εσεί θα αντιμετωπίσετε αυτή την αντίφαση. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο Σβέν Κίγκολτ. Κυρία Λαγκάρτ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα λόγια σας. Είναι καλό που σας βλέπουμε εδώ όπως είπε και ένας από τους προλαλήσατες, ε, σε αυτό τον τομέα των κρυπτονομισμάτων έχουμε τις ε, ε, πολλές πιθανότητες ε, ε, για μια ψηφιακή οικονομία, τι οποίε πρέπει να εξετάσουμε. Οι πολίτες ε, βλέπουν ότι έχουν στη διάθεση τους νέες μεθόδους, έχουν το ίντερνετ, ψηφιακά νομίσματα, μπορούν να έχουν άμεση επιρροή στην διακίνηση των νομισμάτων. Βλέπουμε ότι τα ψηφιακά νομίσματα γίνονται πιο φθηνά και μπαίνουν στα χέρια των του κοινού. Ε, βέβαια, είναι και εργαλείο στα χέρια των εγκληματιών και τα ψηφιακά νομίσματα δεν είναι ε, στα χέρια των ε, διεθνικών επιχειρήσεων. Είναι πραγματικά δυνατό σήμερα κανείς να φέρει σήμερα στην διάθεσή μας ένα ψηφιακό νόμισμα το οποίο θα το εγγυάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ελπίζω ότι θα γίνει. Ευχαριστούμε κύριε Κίκολτ. Ε, ε συνάδελφος ε, Πεντιτσίνη έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, εμείς θα απορρίψουμε την έκθεση αυτή για την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ, γιατί δεν ακούνε οι καλές προθέσεις. Η ΕΚΤ έχει δυστυχώς αποτύχει ως προς την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών ε, και δεν μπορείτε να πείτε ότι φταίει το Brexit για τη μείωση του ΑΕΠ το 18-19 τα μη συμβατικά μέτρα που χρησιμοποιούνται για την επαναχρηματοδότηση των τραπεζών ήταν να διονγκούται το κεφάλαιο των τραπεζών αλλά όχι των νοικοκυριών. Δηλαδή, δυστυχώς, τα παράγωγα των ε, τραπεζών δεν ευεργετούν τις οικογένειες, ε, τα νοικοκυριά και ευθύνεται αποκλειστικά η ΕΚΤ για αυτή τη μεγάλη αποτυχία. Ευχαριστώ. Ας αρχίσουμε το δεύτερο κύκλο με τον Στέφαν Μπέρκερ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε Λαγκάρτε, είναι καλό που ήρθατε σήμερα και μας παρουσιάσατε το νέο στυλ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι θα εξετάσετε τις πολιτικές, θα έχουμε καλύτερη επικοινωνία, καλύτερη επεξήγηση των πολιτικών. Αυτό είναι σωστό και απαραίτητο. Όμως, ε, όταν είναι λάθος η πολιτική, όταν δεν μπορεί να επικοινωνηθεί με άλλο τρόπο, πρέπει κανείς ε, να γίνεται πιο συγκεκριμένος. Έτσι λοιπόν, από την έκθεση βλέπουμε ε, ότι από το 2019 είχαμε 1,9% ε, αύξηση ε, και 2,1% σχέση με το 2020. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν φτάσαμε στο 2% που θέλαμε και τίθεται το ερώτημα το ΙΕΚΤ ε, θα μπει σε μια ε, φάση ε, που δεν μπορεί να βγει. Έχουμε χαμηλούς τόκους, ειδικά στην Γερμανία έχουμε πολύ αρνητικές επιπτώσεις και στις καταθέσεις και στις αποταμιεύσεις και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό πρόβλημα Καλό θα ήταν λοιπόν να δούμε ε, αν μπορείτε να συμπεριλάβετε και στην ε, εξέτασή σας και αυτά τα σημεία. Όπως όσον αφορά τώρα την ε, Τραπεζική Ένωση και την αγγίση των καταθέσεων, είναι πολύ σημαντικό πριν γίνει αυτό να θέσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Δεν κάνουμε ποτέ την ασφάλιση του σπιτιού μας μετά τη φωτιά αλλά πριν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Περέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την παρέμβαση και τον παρεμβατισμό της ΕΚΤ υπό την ηγεσία του Μάριο Τράγκη για να σωθεί η Ευρώπη, να επανορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος και να και για να συνέλθουμε από την γενικότερη χρηματοοικονομική κρίση. Τώρα πνέει ένας νέος άνεμος, από ό,τι φαίνεται, για να ευθυγραμμιστεί η ΕΚΤ με το πράσινο σύμφωνο, σύμφωνο και με την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει όμως να δίνουμε όθηση στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική επιβράδυνση και ύφεση και για να φτάσουμε και στους στόχους του δίκτυ πληθωρισμού. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις που έχουν περιθώρια ελιγμών, δημοσιονομικών ε, ελιγμών και μπορούν να δράσουν πολύ περισσότερο επί του προϋπολογισμού τους. Ευχαριστούμε. Και τώρα έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος ε, Έγκιν Έροκλου. Κυρία Πρόεδρε Λαγκάρτ, ε, κύριε Ντομπρόφσκη, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο της έκθεσης συγκεκριμένα στις αποταμιεύσεις. Μιλήσατε κυρία Λαγκάρτ για το γεγονός ότι θέλετε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα ήθελα παρακαλώ να δω ακριβώ πώς θα συμβεί αυτό γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλο άγχος ως προς την εξαφάνιση των αποταμιεύσεων ε, και φαίνεται ότι οι πολίτες έχουν χάσει την πίστη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επίσης ε, το γεγονός είναι δείγμα της πίστης στην ανεξαρτησία. Επίσης, η ανερντική τόκη, ε, η προστασία, όλα αυτά είναι ζητήματα που επηρέασαν την κατάσταση με τις αποταμιεύσεις. Έχουμε καταθέσει λοιπόν μια τροπολογία ε, που θα τη δείτε στο έγγραφο και με αυτή θέλω να δώσουμε στους πολίτες την εξασφάλιση ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ε, και της πίστης στην ανεξαρτησία θα ενισχυθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αντώνιο Μαρία Ρινάλτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε Λαγκάρτα, διαβάζοντας την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ύφεση η οποία πλήττει την Ευρωζώνη. Δεν νομίζω ότι τα αρνητικά επιτόκια επέτυχαν κάτι. Θεωρώ ότι οι ΜΜΕ επλήγησαν ιδιαίτερα, καθώς και τα νοικοκυριά. Γι' αυτό δεν δόθηκε όθηση πιστοτικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κερδοσκοπία των τραπεζών. Τι θα γίνει με την ποσοτική χαλάρωση που οδήγησε σε μία αύξηση 4,33 αυξάνοντας ε, την νομισματική μάζα τύπου M3 ενώ παράλληλα δεν προωθείται ο αποπληθωρισμός ε, όπως θα έπρεπε. Επίσης προβάλλουμε ε, χρήματα ουρανοκατέβατα, δηλαδή helicopter money, το οποίο δεν είναι ό,τι καλύτερο για την οικονομία μας. Ευχαριστούμε κυρία Φράνσις Φιτσέραλτ. Uh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, κύριε Λακάρτα. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ είπατε ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία στα μέτρα πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πώς θα τα περισσότερο ο κόσμος. Ένα από τα πολύ βασικά θέματα στις εκλογές στην Ιρλανδία ήταν το στεγαστικό έχουν γίνει προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αλλά στο Δουβλίνο, για παράδειγμα, έχουν διπλασιαστεί οι τιμές από το 2010 και η ιδιοκτησία έχει ανέβει 5% από το 2013. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να επικεντρωθείτε περισσότερο στο γεγονό ότι οι τιμέ των κατοικιών αυξάνουν πολύ στην Ευρώπη τελευταία και πολύ γρήγορα και θα πρέπει να υπάρξουν πιο διαφοροποιημένα οικονομικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτό. Ε, έρχομαι και σε κάτι που είπατε εσείς η ίδια πριν γίνεται πρόεδρο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είπατε ότι θα πρέπει έκτη να κατανοήσει και να εξηγεί στον κόσμο, όχι μόνο στις αγορές. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρώπη, τότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πώ θα καταλάβουν οι πολίτε Και πιστεύω ότι αυτό πραγματικά είναι η δημοκρατία πολύ σημαντικό, αλλά πιστεύω επίση ότι το στεγαστικό είναι ζωτική σημασία. Γιατί αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε επαφή με του πολίτε, πρέπει να καταλάβουμε καλά και να λάβουμε υπόψη του τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Οπότε πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Επίγει. Είναι ένα σοβαρό οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα σε πάρα πολλέ χώρε μέλη. Και πιστεύω ότι είναι ένα από τα θέματα που, στα οποία εσεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για να τα κατανοήσει και να προσπαθεί να βρει εναλλακτικέ λύσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Άλφρεντ Σαντ τώρα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον φίλο και συνάδελφο Κώστα Μαυρίδη για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Να επικεντρωθώ και εγώ σε ένα ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκαν και οι προαλήσαντε, αλλά από μια διαφορετική οπτική γωνία. Η κατάσταση των μεγάλων και μικρών τραπεζών στην Ευρωζώνη. Νομίζω ότι υποτιμούμε πόσο δύσκολη έχει γίνει η κατάσταση. Η συζήτηση του ζητήματο αυτού είναι περιορισμένη, γιατί ε, πολλοί θεωρούν ότι αποτελεί μια επίθεση στην ε, πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ιδίω στην διευκολυντική νομισματική πολιτική. Ωστόσο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν πολλέ δυσμενεί συνέπειε, δευτερογενεί συνέπειε και για τι τράπεζε. Έχουμε έναν υπερθεματισμό όσον αφορά τους κανονισμούς που λειτουργεί τελικά αρνητικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα βασίζεται όλο και περισσότερο στον τραπεζικό δανεισμό. Οι τράπεζες λοιπόν καλούνται αυτή τη στιγμή να παρουσιάσουν κερδοφορία, ενώ οι οικονομικές συνθήκες είναι πολλές φορές δυσμενείς. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε κατά αυτόν τον τρόπο πρωταθλητέ στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Νομίζω ότι οι Ευρωπαϊκέ Τράπεζε οι οποίε καλούνται να υποστηρίξουν ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, πολίτε και μικρομεσαίε επιχειρήσει, ενδεχομένω να πληγούν τελικά από την πολιτική που ακολουθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο ζήτησε ο κ. Χάιντερ. Η έκθεση που συζητούμε σήμερα είναι πραγματικά μια. Ε, ε, περιφρόνηση του, του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι ωρεοποιεί τα πράγματα αφενό και απο, αποσιωπά άλλα πράγματα. Το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξη τη ε, Ευρωζώνη παρουσιάζεται ω ε, αποτέλεσμα τη πολιτική χαμηλών ε, επιτοκίων αβάσιμα. Οι απώλειε που οι καταθέτε έχουν υποστεί στην Ευρωζώνη δεν, δεν αναφέρονται καν στην έκθεση. Τα όλο και η μεγαλύτερα ρίσκα, η μεγαλύτεροι κίνδυνοι που διατρέχουν ε, θεσμικοί καταθέτες, όπως για παράδειγμα τα συντοξιακά ταμεία, δεν αναφέρονται καθόλου στην έκθεση. Η, ε, η, δύσκολη, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κεφαλαιαγορές δεν αναφέρονται. Οι κοινωνικές ε, ανισότητε που αυξάνονται λόγω αυτής τη πολιτική δεν αναφέρονται στην έκθεση αυτή. Η, το δημόσιο χρέος που έχει εκτιναχθεί εξαιτίας αυτής της πολιτικής δεν αναφέρεται ούτε αυτό στην έκθεση. Μου, θυμίζουν, μου θυμίζει αυτή η έκθεση τις εκθέσεις που συντάσσονταν στο Ανατολικό Μπλοκ Επικομουνισμού, όπου πάντοτε αναφέρονταν μόνο αυτά που ήθελε η κομματική ηγεσία. Εμείς το γνωρίζουμε αυτό και δεν το δεχόμαστε. Η κυρία Λαλούκ. Κυρία Ραγκάρντ, ευχαριστώ που ήρθατε. Επιλέξατε να συνεχίσετε μια ε, νομισματική πολιτική λεγόμενης νομισματικής ποσοτικής χαλάρωσης και με ανακούφιση πολλοί από εμάς το δεχτήκαμε αυτό γιατί μετά τους εθνικούς ε, εγωισμούς και την κυρίαρχη ιδεολογία στην Ευρώπη δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα πραγματικό προπολογισμό που είναι πράγμα αδιανόητο και απίστευτο για την πρώτη παγκόσμια δύναμη. Αυτή η κατάσταση σας φέρνει αντιμέτωπη εσάς με πολλές ευθύνες και η πολιτική θα πρέπει να είναι υπεύθυνη. Ε, άκουσα πολλά ε, στην ομιλία σας σημεία προόδου, αλλά για την κερδοσκοπία δεν άκουσα. Η ποσοτική χαλάρωση βοήθησε την πραγματική οικονομία και έπρεπε να γίνει, αλλά έφερε και η υπερτροφία ε, αυτής της νομισματικής φούσκας. τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να καταπολεμήσει αυτή την κερδοσκοπία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Παουλ Τάνκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, κυρία Λαγκάχτ. Καταρχάς,